Can we start? αρχίσουμε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Ή μάλλον έχετε έτοιμη την κάρτα ψηφοφορία και, την, και τον κατάλογο ψηφοφοριών. Θα ήθελα να αναπεράσουμε στην έκρηση μερίσιας διάταξης. Όπως γνωρίζετε, σήμερα έχουμε δύο σημαντικές ψηφοφορίε και αναβάλαμε στην επόμενη συνεδρίαση την ψηφοφορία για την έκθεση του συναδέλφου Μαραγκάλ. Συμφωνείτε με την ημέρη σε διάταξη. Ορίστε συνάδελφε. Βέγκερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω την κάρτα ψηφοφορίας μαζί μου. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει λέει ο Πρόεδρος, μπορούμε να περιμένουμε λιγάκι. Και έτσι θα μπορέσετε να την φέρετε. Πάμε στο δεύτερο σημείο έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης τη 7 η Δεκεμβρίου, της προηγούμενης συνεδριάσεως. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Έχουμε διαρμηνία γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, λιθανικά, πολωνικά, σλοβενικά, ουγγαρικά και ρουμανικά παθητικές γλώσσες, ολλανδικά και δανέζικα μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας μέσω web streaming και αποφάσεις των συντονιστών που έγινε στις 11 Ιανουαρίου έχουν αποσταλεί όλα τα μέλη με email στις 12 και θεωρούνται εγκεκριμένα αυτά όταν δεν έχουν αποσταλεί παρατηρήσεις μέχρι τις 14 του μηνός. Ενώ περιμένουμε όλοι να έχετε την κάρτα σας για την ψηφοφορία. Έρχονται με την κάρτα σας τώρα. Πριν ψηφίσουμε λοιπόν, δράτω με τον ως λεπτού της αναμονής να πω. Λοιπόν, έχουμε στις φοφορίες στις τέσσερις. θα έχουμε παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ολλανδικής Προεδρίας με τους δύο υπουργούς παιδείας και πολιτισμού. Διαδοχικά θα τους ακούσουμε πρώτα Λοιπόν, θα έχουμε τη διαδοχή των δύο υπουργών και θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και 5.30. Θα πρέπει σίγουρα να ξεκινήσουμε απαραίτητο συνεδρίες των συντονιστών. Όσον αφορά τις δύο εκθέσεις που θα ψηφίσουμε σήμερα, θα ήθελα να πω κάποια λόγια. Περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές όσον αφορά τη ζωή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν νομίζω ότι η Επιτροπή μας θα μπορεί να το γνωρίσει αυτό το στοιχείο. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα Συμβούλιο Υπουργών σήμερα σημαντικό και πιστεύω ότι είναι προφανές σε όλους ότι χρειάζεται επαναπροώθηση των θεμάτων, των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ενώση, τη παιδεία, του πολιτισμού. Χωρί αυτά δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και εμεί πιστεύουμε ότι σήμερα θα έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση στι διάφορε χώρε και υπάρχει μεγαλύτερη επίγνωση μεταξύ των πολιτών για αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να μπω στην ουσία των αποφάσεων που θα λάβει το Συμβούλιο, αλλά εκφράζω κάποιε σκέψει. Σήμερα μιλάμε για αναστολή του Σέγγεν. Εγώ θα πω μόνο αυτό. Είμαστε στη διεύθερη γενιά των παιδιών του Εράσμου. Τα παιδιά των Εράσμου, εφαντάζονται την Ευρώπη σαν ένα χώρο, χώρο κυκλοφορία, ηθαγένεια, παιδεία, ανταλλαγών και ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι εύκολο να προταθεί να ξανασηκωθούν τα εμπόδια στα σύνορα, να τα προτείνουμε σε αυτή τη γενιά. Θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να μην χαθεί η έννοια της Ένωσης. Δεύτερη παρατήρηση που έχω, την επόμενη Τετάρτη, όπως γνωρίζετε, 27 Ιανουαρίου, είναι η μέρα της μνήμης ε, ανάμνησης της ΣΟΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο πρόεδρος Σούλτς εδώ, πανηγυρικά το έχει αναφέρει εδώ και τρία χρόνια με σταθερή πρωτοβουλία που έχει αναλάβει σε επαφή με τις εβραϊκές κοινότητες, με όλους τους συνομιλητές και επίσημα θα καλέσει το Ευρωκοινοβούλιο όλους εσάς την Τετάρτη στην αίθουσα Μενουχήν 12.45 Τετάρτη 27 Ιανουαρίου. Ήθελα να σας το πω διότι πιστεύω ότι είναι ένα ραντεβού το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Συνάδελφε Βέντα, πρέπει να ξεκινήσουμε. Μπορούσαμε, μπορούμε να λάβουμε υπόψη την ψήφο σα. Γιατί έρχεται η κάρτα σα αλλά δεν έφτασε ακόμα. Καλώ. Πάμε στην πρώτη έκθεση. Έχουμε την γνωμοδότηση. Μα, γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε. Δάμιαν Ντράγκητσι. Όσον αφορά το ενδιαφέρον σχέδιο εκθέσεω Learning EU at School, μάθηση Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολείο, είναι σημαντικό αυτό το θέμα τώρα παρουσιάστηκε στις 12 Νοεμβρίου το σχέδιο κειμένου οι τροπολογίες που ευλέφθηκαν με 19 Νοεμβρίου λάβαμε 228 τροπολογίες πολλές συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, συστάθηκαν ευχαριστούμε τον εισηγητή, τους και τους και τη γραμματεία για όσες προσπάθειε. λοιπόν δεν ξέρω αν θέλει να πει ο συνάδελφο Ντράκιτσι πριν ε, προχωρήσουμε Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, τους κοιόδης συζητητές ε, και τη γραμματεία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη που μου παρίσχουν για την έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς λέει Πρόεδρος, ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Έχετε όλη την κάρτα ψηφοφορίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν συμβαστική τρία του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51 στην επόμενη σελίδα. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 60 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 68 με προφορική τροπολογία. Μαραγάλ. Είστε υπέρ της προφορικής τροπολογίας που συμπεριλαμβάνεται στην τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 του συγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 79 στην 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική α, συνεχίζουμε λέει πρόεδρος τροπολογία 80 Μάιερ υπέρ 88-0 υπέρ ε, κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές ίσως να απορρίπτεται πρέπει να γίνει έλεγχος λοιπόν ξεκινάμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας δεν δουλεύει Εν πάση περιπτώσει απορρίπτεται σαφώς. 19 ψήφοι κατά με 5 ψήφους υπέρ. 82 to reward υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 του συγητού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 107 στην επόμενη σελίδα. Δομινίκ Μπίλτερ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά υπέρ ξανά παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 λέει η πρόεδρος α 119 δεν η πρόεδρος 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πρέπει να γίνει έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 120 120 πέρας απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 ζουλό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 13 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά πρέπει να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 150 αντινόλφη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 μαραγάλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 14 του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 ερ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 167 έλεγχος άρχεται για την 167 πέρας απορρίπτεται Συμβαστική 17 του συγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 έρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 19 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Δεν δουλεύει. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Δεν δουλεύει. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, 11 κατά. 12 κατά. Τροπολογία 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 188 υπέρ, κατά αποχές ίσως να εγκρίνεται αλλά θα ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για την 188 πέρας απορρίπτεται τροπολογία 193 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρινέται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 20 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 208 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ίσως να εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για τη 208 πέρας εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 209 υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 211. Αντινόλφη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίσως να απορρίπτεται, αλλά θέλω να ελέγξουμε. Άρχεται η συμφορία Πέρας. Άλλη μία ψήφος κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 220 υπέρ κατά αποχές ίσως να εγκρίνεται αλλά σε Άρχεται η συμφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 222. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 221. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 223 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται ο έλεγχος πέρας διαφορά. 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Αιτιολογική σκέψη α3. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Γιατί είναι 22 άρχεται η ψηφοφόρια πέρας εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι ταυτόσιμες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 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 του συγγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 με προφορική τροπολογία που συμπεριλαμβάνεται σε ντρόβα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και αναφορά 17, τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία μονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφίσατε όλοι καλώς πέρας ...23 ψήφοι υπέρ, μία αποχή και τέσσερις ψήφοι εναντίον. Συγχαρητήρια στον εισηγητή Δάκητσι Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις για τη δουλειά που έκαναν και τη γραμματεία, δύσκολη δουλειά που έκανα. Και επιτρέψτε μου, για δεύτερη φορά πρέπει να πω έγινε πατέρας μέσα στις γραμματείες. Χθες ή σήμερα το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και ευχαριστούμε για τη δουλειά. Και είσαι ελεύθερος να φύγεις. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη ψηφοφορία. Πάμε στη δική μου έκθεση, στο δικό μου κείμενο για την φτώχεια Ε, Να ευχαριστήσω πολύ τους και όλους και τη γραμματεία για τη βοήθειά τους ε, και ευχαριστώ και τους συμβούλους πολιτικής και τους βοηθούς για τη δουλειά που έκαναν. Είναι μια γνωμοδότηση ενδιαφέρουσα όσον αφορά την ένδια και πώς γίνεται η προοπτική από την πλευρά του φίλου και πλευρά των γυναικών. Ε, γνωρίζετε ότι σαν Επιτροπή Πολιτισμού υιοθετήσαμε Είμαστε μέσα σε αυτό το mainstreaming approach στην προσέγγιση σε όλε τι επιτροπέ, να λαμβάνετε υπόψη αυτή η διάσταση, σε όλε τι πολιτικέ. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το ρόλο και να δούμε και ποιε είναι οι συνθήκε για τι γυναίκε στι διάφορε αρμοδιότητε. Εδώ εστιαζόμεθα στην θηλυκή οπτική γωνία τη φτώχεια και πώ ο ε, αποκλεισμό και η φτώχεια όσον αφορά την στην παιδεία και τη συνεχή κατάρτιση και η φτώχεια, η εκπαιδευτική. Είναι ένα θέμα που αφορά τις γυναίκες που έχουν την αντίθεση αυτή. Έχουν μεγαλύτερο ποσοστό να φτάνουν σε πολλά ψηλά επίπεδα της παιδείας, αλλά ε, ε, υπάρχει και ένα κενό όσον αφορά την αναγνώριση των ποσών του και την καριέρα τους. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι οι δισαγωγή. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε από την παράγραφο 1. Τροπολογία 13 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Jill Evans, χωριστή ψηφοφορία που ζητήθηκε από την Άλντε. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συγγνώμη μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία. Λίγο πιο ήσυχα παρακαλώ. Ευχαριστώ. 18. Υπέρ, κατά, υπέρ, ξανά, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, ψηφίστε. 18. Για τη 18. Πέρασε τις Απορρίπτεται με δύο ψήφους. 19. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ Α, όχι, δεν θα ψηφίσουμε. Είναι απλά γλωσσική φύση η τροπολογία αυτή. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται κατά τμήματα που ζητήθηκε από το άλλο στην 29. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 28? Ωραία, ας ψηφίσουμε για το 28. Παρακαλώ. Πέρασε. Ίσως έκανα λάθος πριν. Με συγχωρείτε. Απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση πάντως. 29. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ για την 37 πέρα στις προφορίες απορρίπτεται για δύο ψήφους 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 κατά τμήματα. Ζήτησε το έλικα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της Για το πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Για τη 47. Πέρασε της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 48. Κατά τμήματα όπως ζήτησε η Άλντε. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ένας ψηφοφορίας πέρας ψηφοφορίας. Για τη συμβαστική 2.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 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές όχι ε, κατά τμήματα όπως ζήτησε η πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ Τέλος σοφορίας για την 72. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1.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 Τέλος της προφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν με 24 υπέρ και 4 κατά. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστήσω και τους σκιώδες συζητητές για το έργο που κάναμε. Προλάβαμε να ψηφίσουμε και εντός του χρονικού πλαισίου που είχαμε θέσει. Uh, Διακόπτουμε για 10 λεπτά διότι καταφθάνει η Ολλανδική Προεδρία σε λίγο. Σε 10 λεπτά λοιπόν στις 4 τα λέμε ξανά.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

Thank

Μπορούμε να ξεκινήσουμε συνάδελφοι, ελπίζουμε να επιστρέψουν και άλλοι συνάδελφοι. Κάναμε μια μικρή υπάψη, μια διακοπή μετά τις ψηφοφορίες. Allora, eh, I, I to, to Italian if me. Θα μιλήσω Ιταλικά αν με επιτρέπετε. Φορές τα ακουστικά σαν έχει την καλοσύνη. Έχω την τιμή να έχω εδώ τον Υπουργό Γέτε Μπούσεμάκα, Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού και Επιστημών, την κυρία Υπουργό, έχει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, σημαντικό, και όπως γνωρίζετε Υπουργέ, είχαμε και άλλη φορά την ευκαιρία να συναντηθούμε δύο φορές. Μία φορά στο Φόρουμ των Νέων, εδώ και κάποιους μήνες, και μετέχαμε και ένα διάλογο πολύ ενδιαφέροντο και εξετίμησα τα μάλα το ενδιαφέρον σας για μια άτυπη συνάντηση πριν την έναξη της Προεδρίας για να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες προτεραιότητες. Πιστεύουμε ήθελα να πω συναδέλφους ότι στη συνάντηση αυτή με την Υπουργό την κυρία Μπουσεμάρκετ και στις 5 παρατέταρτο θα έρθει ο Υπουργός Μάρτιν Φορίν που είναι για την υγεία, επέθυνος για την υγεία και τον αθλητισμό, Υφυπουργός Υγείας και Αθλητισμού. Θα θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας και να σας απευθύνουν και κάποιες ερωτήσεις συνάδελφοι και να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Θα ήθελα να πω ότι είδαμε χαρά ότι οι προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας έχουν επίγνωση ότι περνάμε από δύσκολη περίοδο της ζωής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ελπίζω πραγματικά στο θεματολόγιο των προτεραιοτήτων που έχετε θέσει, αυτά που έχετε θέσει σαν προτεραιότητες στη νέα προώθηση ε, το, της ανώτατης παιδείας και του εκπαιδευτικού συστήματος να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών κατά τη διάρκεια όλης της Προεδρίας. Ζητάμε αυτό και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί Μακρόν γνωρίζουμε ότι η σημαντική ανακοίνωση, ελπίζουμε σύντομα, επί των θεμάτων των δεξιοτήτων και των θέσεων απασχόλησης, skills and jobs, και νομίζω ότι δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα στο πρόγραμμά σας για το 2016 και το νέο θεματολόγιο όσον αφορά την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας θα αποτελέσει αντικείμενο μια κοινή συνεδριάσεως της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Πολιτισμού διότι πιστεύουμε ότι όλη η διαδικασία της κατάρτισης, της απόκτησης δεξιοτήτων της ανώτατης παιδείας και της παιδείας συνδέεται με το θέμα της προσαρμογής των δεξιοτήτων στις νέες ευκαιρίες για εργασία, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και ελπίζω να είναι παρόντες και οι δύο επίτροποι ο... και θα θέλαμε να διαβιβάσουν και στου υπουργού παιδία ή δύο επίτροπε αυτά τα θέματα. παιδεία οι δύο επίτροποι αυτά τα θέματα. Και άλλο σημείο που εντάξατε τι προτεραιοτητε σα είναι η προώθηση τη ηθαγενεια μολι τώρα πριν από λίγο ψηφίσαμε μια έκθεση με τίτλο «Να διδάξουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολείο». Ο συνάδελφος Ντράκητσι ήθελε πράγματι να προωθήσει αυτή την παιδεία ο συνάδελφο ντρακητσι ηθελε αφορά την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, τι κοινέ αξιε το διαπολιτισμικό διάλογο και διαθρησκευτικό, που είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, αλλά επίσης και στη μεσογειακή περιοχή, στην περιοχή της Μεσογείου. Και άλλη μια πτυχή που θεωρώ ότι στηρίζεται είναι ε, το θέμα της αξιοποίησεως της πολιτισμικής κληρονομιάς, της ψηφιοποίησεως αυτής. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που εμείς θέλουμε να προωθήσουμε και το ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε επόμενου μήνε τη προετοιμασία τη μεταρρύθμιση του REFIT, τη αναδιατύπωση τη οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Για τι δημιουργικέ βιομηχανίε, τη δημιουργική βιομηχανία του οπτικοακουστικού τομέα. Θα γίνει διάσκεψη εμπειρογνωμών στο Άμστερνταμ, ότι άκουσα από αυτού. Η νεολαία βεβαίω είναι ένα θέμα το οποίο τη χάνει τη προσοχή και των συναδέλφων, θα χρονοτριβήσω. Θέλω να πω ότι είδαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις σας, τις προτεραιότητές σας και ότι θέλετε να καταλήξουμε σε συγκεντρωμένους στόχους ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Γνωρίζοντας ότι αυτό θα είναι το έτος όπου η Ευρώπη θα κάνει άλμα προς τα εμπρός ή κινδυνεύει πραγματικά να αντιμετωπίσει πολλούς κινδύνους, να το πούμε έτσι. Και αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο και για τις νέες γενιές, κυρίως για τις νέες γενιές. Σας δίνω αμέσω το λόγο για μια εισαγωγή που θα κάνετε και μετά οι συνάδελφοι θα υποβάλουν ερωτήσεις. Ορίστε. Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτέ, πρώτα απ' όλα θέλω να σα ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σα να έρθω εδώ στην Επιτροπή αυτή πολιτισμού. Είναι έτοιμη για μένα που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα τις προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας εκ μέρους του Συμβουλίου. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τις προτεραιότητε της Προεδρίας όσον αφορά την εκπαίδευση και μετά θα αναφερθώ και στις προτεραιότητες μας σχέση με τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωση. Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι δάσκαλοι, οι διευθυντές σχολείων, όσοι ασχολούνται με την πολιτική για την εκπαίδευση έχουν το δύσκολο καθήκον να προετοιμάσουν τους νέους για έναν κόσμο που δεν γνωρίζουμε και για θέσεις απασχόλησης για επαγγέλματα που επίσης δεν γνωρίζουμε. Ένα όμως είναι βέβαιο ότι έχουμε μία αγορά με ελαστικότητα η οποία γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Έχουμε μια σύνθετη κοινωνία που σημαίνει ότι η γνώση δεν φτάνει από μόνη της. Έχουμε ένα κόσμο όπου αντιμετωπίζουμε δύσκολα και περίπλοκα προβλήματα. Όλο και περισσότερο λοιπόν χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να είναι και δημιουργικοί αλλά και να έχουν και πρακτικές λύσεις να προτείνουν. Να υπάρχει ευελιξία και κριτικό πνεύμα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να συνεργαστούν και οι οποίοι να μπορούν να ε, σκεφτούν και να προτείνουν λύση βάσει δημοκρατικών αξιών της ηθαγένειας κάτι το οποίο είναι απαραίτητο σε μια ανθούσα κοινωνία. Είναι πολύ βασικές ε, οι αξίες μας και τα προσόντα των ανθρώπων, τόσο τα γνωστικά όσο και τα μη γνωστικά. Έτσι μόνο μπορούμε να διηγηθούμε σε μια Ευρώπη και τις γνώσεις αλλά και έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις χωρίς αποκλεισμούς. Πολύ σημαντικό όμως είναι να δούμε και τις προκλήσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Ευρώπη πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει ακόμα καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τους πολιτικούς να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις όσον αφορά την αγορά εργασίας. Θέλουμε μια κατάρτιση και εκπαίδευση, η οποία να λαμβάνει υπόψη και να μπορεί να αποφεληθεί από τα προσόντα και τι δεξιοτεχνίε των ανθρώπων. Η Προεδρία μα, ε, λοιπόν, επικεντρώνεται στα εξή και περιμένουμε φυσικά και το Συμβούλιο, της δικές του αντιδράσεις όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πρόσφατα και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δικιά σας Επιτροπή πιο συγκεκριμένα έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον πολυπολιτισμικό διάλογο και στην αγορά εργασίας. Και το Συμβούλιο Υπουργών εξετάζει αυτά τα θέματα και καθορίζει προτεραιότητες για την Ολλανδική Προεδρία. Η προτεραιότητά μας όσον ε, αφορά λοιπόν το εξάμεινό μας είναι οι αξίες, η ριζοσπαστικοποίηση και η μετανάστευση. Θα σας εξηγήσω και τα τρία αυτά. Όσον αφορά λοιπόν τις αξίες, το Συμβούλιο, με το Συμβούλιο συζητάμε πώς θα συνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, όσο γίνεται καλύτερα. Βάσει της νέας ατζέντας της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ολλανδική Προεδρία λοιπόν επ' αυτού οργανώνει δύο συνέδρια. Το πρώτο συνέδριο είναι το Skills for a Lifetime, εξωτεχνίε για μια ζωή. Εδώ λοιπόν κοιτάμε πώς τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να βοηθήσουν για να υπάρξει αυτή η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Για να υπάρχει λοιπόν καλά αυτή η σύνδεση, να γίνει εφικτή, γι' αυτό θα συνεργαστώ και με τον συνάδελφό μου, Άσερ, που είναι υπεύθυνο για τα θέματα εργασίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Συμβούλιο και την προοπτική του Συμβουλίου εκπαίδευση, προκειμένου να συνεργαστούμε καλά για να φτάσουμε σε μια νέα ατζέντα δεξιοτεχνιών. Η δεύτερη διάσκεψη έχει να κάνει με την ανώτατη εκπαίδευση. Εδώ θα συζητήσουμε για τη σχέση ανάμεσα στην ε, ανάπτυξη των δεξιοτεχνιών και τη... μια κοινωνία η οποία αλλάζει συνεχώς και μια αγορά εργασία κυρίω που αλλάζει συνεχώς. Πώς θα εξυγχρονιστούμε, πώς η εκπαίδευσή μα θα εξυγχρονιστεί. Αυτό θα είναι κεντρικό σημείο. Δεύτερη προτεραιότητα τώρα για την Ολλανδική Προεδρία είναι η ριζοσπαστικοποίηση. Ιδιαίτερα μετά τις φρικτές πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι είναι ζωτική σημασία η ριζοσπαστικοποίηση και η αναγνώριση συνέπειές της να είναι πράγματα τα οποία θα προσέξουν τα σχολεία και οι καθηγητές. Στο Συμβούλιο λοιπόν για τη συζήτηση θα λάβουμε υπόψη μας διάφορα από την δήλωση του Μαρτίου που μας πέρασε στο Παρίσι. Και αυτά είναι η εκπαίδευση, η αγωγή του πολίτη δηλαδή, η ενίσχυση του ρόλου του δασκάλου και τα μέσα ενημέρωσης. Θέλουμε τις βέλτιστες πρακτικές να τις ανταλλάξουμε μεταξύ μας σε αυτά τα πλαίσια βάσει αυτών των τριών θεμάτων. Στόχος μου λοιπόν είναι οι χώρες μέλη να αποκτήσουν αυτή την όθηση για να προωθήσουν τα όσα αναφέρει η δήλωση του Παρισιού. Και αυτό ακριβώ νομίζω ότι στήσατε και εσείς στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα όταν αναφερθήκατε στον διαπολιτισμικό διάλογο και την εκπαίδευση. Η τελευταία προτεραιότητα είναι η μετανάστευση. Και εδώ το Συμβούλιο Εκπαίδευσης Πολιτισμού και Αθλητισμού θα δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα για να βρεθούν οι σωστές λύσεις όσον αφορά την ροή προσφύγων και πώς αυτοί θα ενταχθούν στην εκπαίδευση. Στο τελευταίο τέτοιο συμβούλιο η Λουξεμβουριανή Προεδρία ήδη είχε τεθεί το θέμα. Δεδομένων όμως των εξελίξεων είναι πολύ σημαντικό να το ξαναδούμε και να ανταλλάξουμε και πάλι εμπειρίες μεταξύ μας από αυτού. Δεν πρέπει εδώ να ξεχνάμε ότι η κοινωνική ένταξη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαι πεπισμένη ότι μεταξύ των μεταναστών μας είναι πολλοί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολλά στις κοινωνίες μας και στην Ευρώπη ολόκληρη. Κυρίες και κύριοι, προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας πάνω στα θέματα αυτά. Εδώ λοιπόν ε, σταματάω με την εκπαίδευση και θα περάσω στις προτεραιότητές μας όσον αφορά τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης. Ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, τα οπτικοακουστικά μέσα είναι πράγματα πολύ σημαντικά και είναι πράγματα τα οποία μας ενώνουν μέσα στην Ευρώπη. Συγχρόνως όμως είναι αυτά που μας βοηθούν να καταλάβουμε, να ακούσουμε, να δούμε και να αισθανθούμε και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας. Μέσα λοιπόν σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, μια Ευρώπη της γνώσης, είναι πολύ σημαντικό να έχουν πρόσβαση στα αγαθά αυτά όλοι όσοι κατοικούν στην Ευρώπη. Πέρα συνόρων. Για τον πολιτισμό λοιπόν η Ολλανδική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στις εκπομπές online και στο οπτικοστικό περιεχόμενο. Τον Ιούνιο οργανώνουμε μία διάσκεψη για την ψηφιοποίηση των πολιτισμικών ε, συλλογών. Στο Άμστερνταμ θα γίνει η διάσκεψη αυτή και θα χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα από αυτήν την διάσκεψη και στο Συμβούλιο όπου θα συζητήσουμε στις 31 Μαΐου. Το Συμβούλιο θα δώσει ιδιαίτερη σημασία βέβαια και στο Ευρωπαϊκό είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο για την ψηφιακή μας κληρονομιά. Η Ευρωπαϊκή συνδέει ήδη 45 εκατομμύρια αντικείμενα από πάνω από 3.000 αρχεία, μουσεία και βιβλιοθήκες. Ένα σωρό επαγγελματίε από ολόκληρη την Ευρώπη έχουν συμμετάσχει στο έργο αυτό και μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όμως τώρα είμαστε μπροστά στην επόμενη πρόκληση. Και αυτή είναι πόσο θα φτάσουμε σε ένα ευρύ κοινό πώς θα μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή. Πολύ ωραίες ψηφιακές συλλογές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κόσμο. Τα πειραματικά προγράμματα υπάρχουν ήδη και έχουν να κάνουν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην εκπαίδευση. Στο Συμβούλιο λοιπόν ως πρώτη μου φιλοδοξία έχω να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό η συμμετοχή των χωρών μελών, γιατί το Ίδρυμα Ευρωπαϊκό δεν μπορεί να τα κάνει όλα από μόνο του. Χρειάζεται και εθνική πολιτική κατάλληλη για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και συμμετοχή όλων των χωρών για να μπορέσει να προχωρήσει το σχέδιο αυτό. Και τρίτον, πρέπει να δούμε το θέμα της χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό εξαρτάται από χρήματα κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από εθελοντικές προσφορές από τις χώρες μέλη. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο Συμβούλιο σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά για μια πιο μόνιμη χρηματοδότηση. Ελπίζω επίσης ότι θα συμφωνήσει το Συμβούλιο στις 31 Μαΐου επ' αυτού. Και χαίρομαι που ο Επίτροπος Ούτιγκερ επίσης εξέφρασε τον ενδιαφέρον του για το θέμα αυτό. Σήμερα ήρθα για να ακούσω και τη δικιά σας γνώμη για το Ευρωπαϊκό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάρα πολύ θετικό από την αρχή όσον αφορά το σχέδιο αυτό του Ευρωπαϊκού και ελπίζω ότι η συμμετοχή σας αυτή στο Ευρωπαϊκό θα συνεχιστεί. Κυρίε και κύριοι, έτσι έρχομαι στη δεύτερη προτεραιότητα που είναι τα οπτικοακουστικά. Ποια είναι τα σχέδια της Προεδρίας επ' αυτών. Όπως και εσείς, το Συμβούλιο περιμένει πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας όσον αφορά τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Την άνοιξη, κατά πάσα πιθανότητα. Στο μεταξύ, κάνουμε συζητήσεις για αυτά τα θέματα, όπως την αναθεώρηση όσον αφορά τα δικαιώματα των δημιουργών, και γενικότερα την ε, πολιτική μας όσον αφορά την ε, ψηφιακή αγορά. Επίσης οργανώνουμε μια διάσκεψη για το οπτικουστικά στο Άμστερνταμ. Τα αποτελέσματα της διάσκεψης αυτής θα συζητηθούν μεταξύ των Υπουργών στο Συμβούλιο. Θέλουμε να υπάρχει ανταλλαγή των ε, έργων αυτών των οπτικουστικών και πέρα των συνόρων. Επίσης, διάδοση των έργων σε ολόκληρη την Ευρώπη, είτε πρόκειται για ταινίε, είτε πρόκειται για ντοκιουμαντέρ ή κινούμενα σχέδια, οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η ψηφιακή επανάσταση παίρνει μια νέα διάσταση. Κυρίως επειδή χρησιμοποιείται τόσο πολύ από τις νέες γενιές. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους φορείς και τους παραγωγούς, το βίντεο on demand για παράδειγμα ή τα κοινωνικά μέσα έχουν αλλάξει πάρα πολύ το ψηφιακό τοπίο. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε νέες στρατηγικές. Και εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε επικριτικοί όσον αφορά τις πολιτικές μας και τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Τέλος. για τις ε, συζητήσεις, διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Ό,τι όμως και να γίνει, όσο και αν προχωρήσουμε ή δεν προχωρήσουμε, όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει ο πολιτισμός και τα μέσα ενημέρωσης. Και όχι μόνο για την οικονομία και την απασχόληση. Πρόκειται για το ίδιο το πρόσωπο, τη φωνή και την καρδιά που χτυπάει μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Ευρώπης. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι αυτές οι σκέψεις θα μας καθοδηγήσουν και στο έργο μας στο μέλλον. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και σας για τη βοήθειά σας. Κυρίες και κύριοι, προσβλέπω στην σημερινή ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, όπως επίσης προσβλέπω και σε καλή συνεργασία μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you so much for your intervention. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και για τις προτάσεις που κάνατε. Αυτά που είπατε ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας επιστησίες και την προσοχή που δίδουμε. Εξάλλου, αναφερθήκατε σε κάποια ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενα σημαντικών εκθέσεων που συνέταξε αυτή η Επιτροπή ε, και έκανε διοργάνωση ακρόαση από αυτόν ή ανέθεσε έρευνε. Η πρώτη ήταν για την ποικιλομορφία και τον πολιτισμικό διάλογο, το θέμα της ηθαγένειας, της παιδείας, ε, των νέων στην Ευρώπη και τα άλλα θέματα που μας ενδιαφέρουν για τον πολιτισμό. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ πολιτισμικού περιεχομένου, μεγαλύτερη πρόσβαση στη δημιουργικότητα και στον πολιτισμό και τη νέα ψηφιακή πρόκληση. Γι' αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και μιας ε, σημαντικής εκθέσεως που εγκρίναμε στο Σασβούργο στην προηγούμενη Ολομέλεια ακριβώς με μεγάλη παρουσία του εισηγητού σε αυτό το θέμα και ασχολούμεθα και με το θέμα των μεταναστών. Θα κάνουμε και ε, ακρόαση όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών και κάναμε και μια ημερίδα, ένα εργαστήριο όσον αφορά την πρόληψη της ρίζοσπαστικοποίησης, ρίζοσπαστικοποίησης συγγνώμη. και το θέμα του εξυγχρονισμού της ανώτατης εκπαίδευσης να μπορεί να εντάσσονται όλοι είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Δίνω το λόγο στους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Τρία λεπτά παρακαλώ στους συντονιστές των ομάδων και δύο λεπτά για τα άλλα μέλη για να προλάβουμε το χρόνο. Φεράιαν Καμερέβερ Τρούπελ είναι οι πρώτοι που ζήτησαν το λόγο και μετά διακόνου. Φεράιαν. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε μαζί μας εδώ σήμερα και που μας μιλήσατε για τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Αναφερθήκατε σε σημεία που συζητούμε κι εμείς και που βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και των εκθέσεων μας. Θα ήθελα όμως να μας δώσετε κάποιες πιο λεπτομερείς ε, πληροφορίες από τη δική σας πλευρά για αυτά τα σημαντικά θέματα, διότι ε, πρόκειται για θέματα όπου και εμείς ε, θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε, θα μπορούσαμε να ε, συνεισφέρουμε και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολλά από αυτά επίσης αποτελούν αρμοδιότητες των εθνικών κρατών και ακριβώς λόγω της μεγάλης ε, ευρύτητας του ζητήματος, ε, της ενσωμάτωσης, ε, της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτά τα θέματα είναι κυρίως εθνικά θέματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν πώς μπορείτε εσείς να παρακινήσετε τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση γιατί τα κράτη-μέλη έως τώρα έχουν επιδείξει μάλλον μικρό επίπεδο προθυμίας να δραστηριοποιηθούν. Θεωρώ επίσης ότι είναι θετικό το γεγονός ότι στον τομέα της ε, απασχόλησης των νέων και της εκπαίδευσης είναι σημαντικό να κοιτάξουμε ποιες είναι οι βασικές επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτεί ή που χρειάζεται η αγορά εργασίας αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανατραπούν ε, οι παραδοσιακές αξίες ε, όσον αφορά τις ε, βασικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, συντάξαμε και μια έκθεση για το πώς διδάσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο της Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται τη συνδρομή και των κρατών μελών. Υπάρχει κάποια ε, δική σας στόχευση στο συγκεκριμένο τομέα, διότι ε, αντιμετωπίζουμε και τον κίνδυνο ε, μιας κάποιας διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υποτίμησης της αξίας των ε, ευρωπαϊκών αξιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπάρχει κάποιο σχέδιο από τη δική σας πλευρά για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί ε, η ευαισθητοποίηση γύρω από, ε, γύρω ευρωπαϊκά ζητήματα. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκά, ε, χαίρομαι πολύ που εκφράσατε την στήριξή σας στο πρόγραμμα αυτό. Εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε εκφράσει και τα προηγούμενα χρόνια την υποστήριξή μας για το πρόγραμμα αυτό, κάτι που δεν ήταν πάντοτε εύκολο, ιδιαίτερα και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, διότι πολύ συχνά ακούμε το αντεπιχείρημα ότι ο πολιτισμός αποτελεί εθνική αρμοδιότητα ε, και γι' αυτό το λόγο δεν, ε, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να δοθεί χρηματοδότηση από ευρωπαϊκή πλευρά στον πολιτισμό, αλλά εγώ σε κάθε περίπτωση χαίρομαι για το γεγονός ότι εκφράσατε την υποστήριξή σας προς μια τέτοια κατεύθυνση εκ μέρους του Συμβουλίου. Για τους σοσιαλιστές. Η κυρία Κάμερβερτ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ για να μας προσέσετε τις προτεραιότητες σας για το εξάμεινο της δικής σας προεδρίας. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε όλα τα σημεία που αναφερθήκατε, γιατί ήταν ευρύτατα. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Αναδείξατε ότι ο πολιτισμός και τα μίντια είναι απαραίτητο στοιχείο για την λειτουργία της δημοκρατίας μας και δεν θα πρέπει να εξετάζονται απλά και μόνο ως εμπορεύματα, διότι είναι πολύ περισσότερο από αυτά. Είναι απαραίτητο στατικό στοιχείο της δημοκρατίας και θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό και να σας παρακαλέσω το μέτρο των δυνατοτήτων σας βεβαίως να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα και στο Συμβούλιο διότι διαρκώς διαπιστώνουμε ότι αναλόγως με, το, με ποιον μιλά κανείς στο Συμβούλιο για παράδειγμα με υπουργού ε, βιομηχανίας ή οικονομίας αυτό το στοιχείο ε, μάλλον ξεχνιέται και πολύ περισσότερο τονίζεται η οικονομιας αυτο το στοιχειο μαλλον ξεχνιεται διάσταση του πολιτισμού χωρίς να λαμβάνεται επαρκώς ε, υπόψη η σημασία που έχουν τα μίντια και ο πολιτισμός για την ποικιλομορφία και την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ε, ελπίζω κάποια στιγμή ίσως όχι στη δική σας προεδρία, αλλά σίγουρα φέτος να συζητήσουμε για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα και θα πρέπει αυτή τη διάσταση που μόλις ανέφερα ε, να μην την ξεχάσουμε, να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στην οικονομική σύγκληση, αλλά και στη σύγκληση ε, όσον αφορά τον πολιτισμό. Κάτι ακόμη. Γνωρίζετε ότι ως Επιτροπή έχουμε τονίσει σε πολλές εκθέσεις μας ότι θα θέλαμε το 2018 να χαρακτηριστεί ως έτος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι στο Συμβούλιο υποστηρίζουν μια τέτοια προοπτική γιατί ένα τέτοιο έτος θα είχε σημαντικότατες θετικές επιπτώσεις και στην οικονομία και στον τουρισμό και στην ανάπτυξη της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θεωρούμε ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συνεισφέρει και στην οικονομία. Αφετέρου, ωστόσο, ακούμε ότι η διάθεση ε, ε, στην Κομισιόν δεν είναι ιδιαίτερα θετική απέναντι σε μια τέτοια ε, προοπτική να οριστεί το 2018 ως έτος πολιτιστικής κληρονομιάς γιατί θεωρείται από εκείνη την πλευρά ότι δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα αυτό στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Εμείς φυσικά διαφωνούμε με αυτό και θα θέλαμε να λάβουμε υποστήριξη ε, από το Συμβούλιο να αποφασίσει το Συμβούλιο δηλαδή να χαρακτηρίσει το 2018 ως έτος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς. Θα μας βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ Πέτρα. Έλκα Τρούπελ τώρα. Σε μινούτη. Τρία λεπτά. Ehm, yes, thank you very much for... Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία ε, και που είστε εδώ ε, για να μιλήσουμε. Μια ερώτηση έχω για το Ευρωπαϊκό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το πρόγραμμα και είχαμε και δυο μεγάλες εκθέσεις ε, συντάξει. Ε, θα ήθελα να βρούμε τρόπο χρηματοδότησης του Πεάνα όχι μόνο σε ετήσιο επίπεδο αλλά και μακροπρόθεσμα ως πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να ε, αναδείξουμε ότι μας ενδιαφέρει να χρηματοδοτηθεί το Ευρωπαϊκά από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ε, αντικείμενο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολιτού ε, δημοσιονομικού πλησίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες φήμες προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκά πρέπει να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Για το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Έχουμε διοργανώσει και κάποιες δημόσιες ακροάσεις και ακούσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει θρησκευτική εκπαίδευση στα σχολεία χωρίς να περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένα δόγματα. Θα πρέπει οι μαθητές δηλαδή να γνωρίζουν διάφορες πληροφορίες για τις διάφορες θρησκείες και έχουμε διαπιστώσει μέσω μελετών και μέσω γυναικών της μουσουλμανικής κοινότητας ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τον εντοπισμό διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης και ότι χρειάζονται πολύ ε, σημαντικές πληροφορίες και γνώσεις για την ευρεία ερμηνεία του Κορανίου, γιατί οι σαλαφιστές κάνουν το αντίθετο, έχουν, ε, εφαρμόζουν μια στενή ερμηνεία του Κορανίου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, πιστεύω, περισσότερα προγράμματα, περισσότερη χρηματοδότηση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες να παρεμβαίνουν στην υπέρ της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και θα ήθελα να μας πείτε εσείς τι σκοπό έχετε ως Ολλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ, συνάδελφος Διακόνου. Έχει το λόγο. Ζανοδιέσκη και μετά διακόνο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που μπορώ να σα καλωσορίσω σήμερα. Έχω τρει ερωτήσει. Η πρώτη, πρόσφατα σαν Υπουργό Πολιτισμού επί Πολωνικής Προεδρίας θυμάμαι ότι είχαμε την ευκαιρία να προωθήσουμε, να προωθήσει κανείς τη χώρα του κατά διάρκεια του εξαμήνου. Σας είναι υπουργό. Χρησιμοποιείτε αυτή, θα χρησιμοποιήσετε δυνατότητα να προωθήσετε την Ολλανδία στον πολιτισμικό τομέα. Δεύτερον, θυμάμαι ότι η χώρα σας προετών έκανε σοβαρές περικοπές όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού. Η Προεδρία σας δίνει την ευκαιρία να αυξήσει τη χρηματοδότηση που θα διατίθεται στη χώρα σας. Τρίτη ερώτηση. Για την συνέχιση των στατιστικών στοιχείων. Τη συνέχεια των στατιστικών δεδομένων και ποια χρήση κάνετε. Στατιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν την οικονομική αξία ε, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κλπ. κλπ. Τέταρτο σημείο. Αντίθετα με αυτά που είπατε, η Ευρωπαϊκή χρειάζεται διαφήμιση, πρόθεση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αυτοπροθυθεί ε, σχεδιάζετε κάποιες εκστρατείες για να προωθήσετε την Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Διακόνου και μετά η Τζουλι Ward. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Καταρχάς θα προσπαθήσω, θα ήθελα να σας συγχαρώ. Θα είμαι πολύ σύντομος είναι, θα είμαι σύντομο, σπάνιο για έναν πολιτικό. Αναφερθήκατε σε όλα τα θέματα που μας αφορούν και εμά. Μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Έτος της Κληρονομιάς, ε, την Ευρωπαϊάνα. Θα ήθελα όμως να πω κάτι παρόλα αυτά. Δεν αμφισβητώ ότι διαπιστώσατε ότι για να καταπολεμηθεί η ρίζοσπαστικοποίηση και όλα αυτά που συνεπάγεται για τη μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών Τα όπλα, οι πληροφορίες δεν αρκούν. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη ριζοστατικοποίηση χάρη στις ευρωπαϊκές αξίες και να προωθούμε τις ευρωπαϊκές αξίες όπως προωθούμε και άλλα μέσα για να υπερασπιστούμε. Ένα λεπτό και μόνο κάνατε, είσαι συντομότατος. Evans, συνάδελφε Evans, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Χαίρομαι που τονίσατε την παιδεία. Εγκρίναμε μια πολύ καλή έκθεση το απόγευμα όσον αφορά τη σημασία που έχει εκπαίδευση για να καταπολεμήσει την φτώχεια και να εξισορροπήσει την κατάσταση των δύο φύλων. Ε, για διάφορα θέματα που θίξατε, βλέπω ότι υπάρχει μια κοινή ανάγκη. Η ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, της οργανώσεως των, της κοινωνίας των πολιτών. Και για να πλησιάσουμε τον κόσμο πρέπει να τον πλησιάσουμε στη γλώσσα του. Καμιά φορά στην... κυριολεκτικά. Εκπροσωπώ την Ουαλία που είναι δίγλωση. Είχαμε εκθέσεις της Επιτροπής κατά παρελθόν για τις μειονοτικές γλώσσες και τις μειονοτικές, ε, το μειονοτικό πολιτισμό και πρέπει να, τι πρέπει να υποστηριχθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο παράγων Πώς θα το προσεγγίσετε αυτό το θέμα υπό την Προεδρία σας. Julie Βόρτ, συγγνώμη. Είχαμε άλλη εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου που θα μιλούσε πριν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε- επίσης που αναφερθήκατε εκτενώς στην έκθεση για το διαπολιτισμικό διάλογο. Ήμουν η βασική συγγήτρια και ενεκρίθη χωρίς τροπολογίες με μεγάλη πλειοψηφία την περασμένη εβδομάδα. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω ότι επέλεξα την έκθεση βλέποντας με πολύ θετικό μάτι τους νέους και το δυναμικό που μας προσφέρουν. Προσφέρουν στην κοινωνία μας, επιλύουν τα προβλήματα, ξέρουν περισσότερο από τους άλλους πώς να ζουν μαζί, δεν έχουν γεννηθεί με μυσαλλοδοξία. Το Σαββατοκύριακο στη Βορειοδυτική Αγγλία ήμουν παρούσα στο Youthphoria. είναι ένα κοινοβούλιο των νέων, μια μορφή τέτοια, και επέλεξαν για την εκστρατεία τους μια εκστρατεία με τίτλο «Εκπαίδευσε και μην μισείς». Αυτός είναι ο τίτλος. Ενδιαφέρονται και θέλουν εκεί επίσημη και ανεπίσημη παιδεία θεωρούν ότι μπορεί να τους δώσει μια βάση, μια πλατφόρμα για να προσπαθήσουν να είναι ε, πιο ε, φιλικοί προς τους άλλους διότι έχουν διαφορετικό υπόβαθρο εθνοτικό αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι νέοι και ενδιαφέρονται πολύ και για το μίσος που στρέφεται κατά των ατόμων με αναπηρίες κατά τον ΛΟΑΔ και τον εργάζεται κανείς στην επίσημη παιδεία είναι ένας τρόπος για να αντιταχθεί σε όλα αυτά τα φαινόμενα επιτυχώς. Συνάδελφε Χιμένες Μπαμπάτ, καλωσορίζουμε και τον Υπουργό Και εγώ συγχαίρω την ε, Ολλανδέζα Υπουργό Πολιτισμού και Εκπαίδευσης για το Ευρωπαϊάνο πέρα των άλλων που με ενδιαφέρει εμένα όλος ιδιαίτερος. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν ευρωπαϊκό λόγο κοινό ο οποίος να σφυριλατεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Άκουσα και το σχόλιο της κυρίας Τρούπελ Πώς να συμφιλιώσουμε λοιπόν τις διάφορες ιστορίες αυτές ε, πολιτιστικές και ιστορικές που έτσι καλώς είναι δύσκολο να συμφιλειωθούν στην Ευρώπη από τα παλιά έθνη. Πώς να τα συμφιλιώσουμε αυτά με τους νέους που μας έρχονται στην Ευρώπη, μετανάστες, πρόσφυγες και τα που συνοδεύονται από τη δικιά τους βέβαια ιστορία, που είναι διαφορετική. Συνάδελφοι Σοϊντρόβα, μία από τις τέσσερις αντιπροέδρους της Επιτροπής Πολιτισμού σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Γνωρίζω ότι το σύστημα το εκπαιδευτικό της Ολλανδίας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ καλό ιστορικό στον αφορά την ένταξη ε, και την καινοτομία. Ελπίζω ότι η δική σας ε, Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη σημασία που έχει η παιδεία Αναφερθήκατε σε κάποιες πτυχές που θέλετε να τονίσετε. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια θέματα θα τα θέσετε σαν θέματα διασκέψεων και πώς επίμαχα θα είναι τα θέματα. Η μετανάστευση θα είναι κάτι επίμαχο, η ριζοσπαστικοποίηση θα είναι επίμαχο θέμα. Θα είναι δύσκολο να επιμένετε, να επιμένετε τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερη προσοχή σε αυτά. Αλλά θα ήθελα να, ενθαρρύνω, να σας ενθαρρύνω να δώσετε τη δέουσα προσοχή και να χρησιμοποιήσετε και τις εκθέσεις βέβαια της Επιτροπής μας. Και δεύτερον, η Ευρωπαίνα, Θα ήθελα να πω ότι ο Τσέχος Υπουργό Πολιτισμού θα σας στηρίξει 100%. Μπορείτε να βασίζεστε στην πλήρη υποστήριξη της τεχικής δημοκρατίας διότι θεωρούμε ότι η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς είναι ένα έξοχο πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει η ευρωπαϊκή κληρονομιά να γίνει πιο ορατή. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Κέστερ. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Χάρηκα ιδιαίτερα που ως στόχο του έργου σας τονίσατε τον στόχο μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας γιατί είναι σημαντικό να υπάρξουν συμμετοχικές διαδικασίες γιατί και στο θέμα των προσφύγων το ζητούμενο δεν είναι μόνο να, να προσαρμοστούν αλλά πώς θα μπορέσουν οι ίδιοι να συμμετάσχουν στις κοινωνικές δραστηριότητες και εδώ η εκπαίδευση και ο πολιτισμός έχουν να ε, διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από τεράστιες ανισότητες. Εσείς αυτό το εξάμεινο που θα έχετε την Προεδρία δεν θα μπορούσατε να εξετάσετε με ποιον τρόπο η εκπαίδευση θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε πολλές χώρες οι άνθρωποι που μειονεκτούν κοινωνικά, μειονεκτούν και στον τομέα της εκπαίδευσης. Και αν δείτε και τους τρομοκράτες, συνήθως πρόκειται για ανθρώπους που ήταν φτωχοί ή που είχαν χαμηλή συμμετοχή σε πολιτικές και κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτό είναι το ένα. Ε, ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να τονίσω είναι, ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η έννοια της διαβίου μάθησης, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο του ομιλητή. Sorry. Das endet oft die Eurostat. Ε, ένα δευτερόλεπτο λέει η Πρόεδρος. Πολλές φορές η, τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat γύρω από τη διαβίου μάθηση αφορούν ηλικιακές ομάδες έως την ηλικία των 60. Ωστόσο, η διαβίωμα θα έπρεπε να υπερβαίνει πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο όριο των 60 ετών. Μοργάνο, ευχαριστώ Υπουργέ. Στην εισαγωγή σα αναφερθήκατε σε δύο διασκέψει: Μία για το θεματολόγιο των δεξιοτήτων και το άλλο για την εκπαίδευση, για ανώτερη ικανότητα εκπαίδευση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω θετικά να στηρίξω αυτά που είπατε, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποιε είναι οι αρμοδιότητε τη Ενώση όσον αφορά αυτά τα θέματα. Αλλά αν δεν πλησιάσουμε ένα τον άλλον, όπω κάνουμε στην Επιτροπή και ανταλλάσσονται καλέ ε, πρακτικέ, δεν θα κάνουμε βήματα πρόοδο Και το λέω αναφερόμενο στο ρόλο που παρόλα αυτά μπορούν να παίξουν αυτέ οι επιλογέ σε σχέση με την κοινωνική ένταξη. Δεύτερο, τονίσατε το διαπολιτισμικό διάλογο. Θεωρώ ότι αντικειμενικά είναι η επιλογή ε, που είναι απαρέκλητη και με αναφορά στη διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ του θέματος του διαπολιτισμικού διαλόγου από τη μια και των προτεραιοτήτων από την άλλη πλευρά που αναφέρατε για την Ευρωπαϊκή. Είναι σαφές ότι ένας διάλογος διαπολιτισμικό υπάρχει όταν υπάρχουν θέσει, όταν υπάρχουν ταυτότητε που συζητούν. Και εν αυτή τη ενία συμμερίζομαι διάφορε παρατηρήσει των συναδέλφων, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημείο αδυναμία που τονίσατε. Δηλαδή τη, την σχετική χρήση του τεράστιου υλικού που έχουμε ε, έναντι διαφόρων επιλογών που θα μπορούμε να κάνουμε. Πόσο καλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαθέσιμο υλικό. Μετά η συνάδελφο Πέτρα αναφέρθηκε σε κάτι και θα ήθελα να το τονίσω κι εγώ. Δηλαδή ότι το 2018 θα πρέπει να γίνει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού Γνωρίζουμε ποια είναι η θέση που εκφράστηκε στο Συμβούλιο. Υπάρχει ισχυρή υποστήριξη. Χρειάζεται ανάγκη, υπάρχει ανάγκη να επιμείνουμε και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπούλ. Thank you, uh, Chairman. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, η Επιτροπή πολύ συχνά ζητά να γίνονται εξατίες στην Ευρώπη για να προωθούνται τα ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση. Ψηφίσαμε και μια έκθεση σχετική ε, το απόγευμα μια έκθεση με θέμα να μαθαίνουμε την Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία. Αποκλείεται ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο δημοψήφισμα για το Βρετανική έξοδο, το Brexit, μέσω εκστατιών στα μέσα ενημέρωσης, μέχρι να διεξαχθεί το δημοψήφισμα θα γίνει, το αποκλείεται και αν γίνει, ε, τι μπορεί να παραχθεί και τι μπορεί να διανεμηθεί αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. Ο κ. Γραμματικάκης. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Εγώ χάρηκα γιατί η υπουργό ήταν πολύ σύντομη και περιέλαβε όλα τα σπουδαία ζητήματα. Βέβαια είμαι πάλι βέβαιος ότι η θέληση της Προεδρίας θα είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα γιατί παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής Πολιτισμού και ειδικά της Προέδρου νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο αισθάνεται την αξία του πολιτισμού λίγο τη συμμερίζεται. Όπως εσείς κυρία Υπουργέ και δύο ερωτήσεις πολύ γρήγορες. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων που εκκρεμεί. Έχετε κάποιες δικές σας απόψεις γιατί όπως είπατε κατά το Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κανείς δεν ξέρει με την κατάσταση που υπάρχει θα έρθει η νομοθεσία. Και δεύτερο, τα πολύ πετυχημένα προγράμματα αυτής της Επιτροπής. Να αναφέρω για πολλωστή φορά το έρασμος. Έχουν πολλαπλές δυσκολίες. Έχετε στο μυαλό σας κάτι να τα διευκολύνετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Όπως βλέπετε κυρία Υπουργέ, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την Ολλανδική Προεδρία. Θα σας δώσω πολύ ευχαριστώ λοιπόν το λόγο διότι πιστεύω ότι ετέθησαν πολλές απαντήσεις, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσετε σε όλες, αλλά ίσως μπορεί να τις ομαδοποιήσετε κάπως και να προσπαθήσετε να απαντήσετε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε ήδη βέβαια εδώ και τον Υπουργό του Κιφανρή, οπότε θα πρέπει μέσα σε 10 λεπτά να ολοκληρώσουμε, αν έχει την καλοσύνη αυτή την συνάντησή μας. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι, πολλές ήταν οι ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω όντως να συγκεντρώσω κάπως τις ερωτήσεις σας για να απαντήσω μαζί σε πολλές. Πολλοί από σας αναφερθήκατε στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι εκείνη η οποία θα προετοιμάσει τις νέες γενιές για να τα καταφέρουν με υπευθυνότητα είναι ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπη η εκπαίδευση, όπως είπε και ο κύριος Κίστερ, πράγματι και για να καταπολεμήσει τις κοινωνικές ανισότητες. Γι' αυτό και έχουμε την κατάλληλη πολιτική. Έχουμε το Education and Training Monitor. Και στο Συμβούλιο θα φροντίσουμε να περάσει το σωστό μήνυμα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όντω λοιπόν η εκπαίδευση και ο πολιτισμό είναι ζωτική σημασία προκειμένου η Ευρώπη να μην είναι μόνο βιομηχανική πολιτική, όπω είπε και η κυρία Κάμερβελτ, αλλά να πρόκειται για τι αξίε, για τι αρχέ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει κοινωνικό διάλογο. Εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί ακριβώ εδώ είναι που έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορούμε πολλά να πούμε για την εκπαίδευση, να αναρωτηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψει να συνομιλήσουμε και έρχομαι στο Erasmus Συν, που είναι όντως ένας τρόπος για να προωθήσουμε τον κοινωνικό διάλογο και την πολυπολιτισμικότητα, προκειμένου οι νέοι να μάθουν τι είναι αυτό που απασχολεί τους άλλους. Να μάθουν τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και άλλες χώρες επίσης έτσι έχουν να μάθουν από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς οργανώνουμε, πολύ σωστά με ρωτήσατε, τι μέσα έχουμε για να πετύχουμε αυτούς τους τόσο ωραίους στόχους. Έχουμε λοιπόν το Erasmus αλλά έχουμε και τη συνεργασία με τον ανοιχτό συντονισμό, με τη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού και έχουμε και το e ΙΤ 2020 που θα αναφερθεί τον Αύριο και στο Συμβούλιο Έχουμε και πολιτικές που μπορεί να μην είναι δεσμευτικές, υποχρεωτικές, αλλά όσο να οι χώρες μέλη ενημερώνονται και τις προωθούν. Για την κυρία Ζετρόβα θέλω να πω ότι στο Συμβούλιο πράγματι πρέπει να κάνουμε και τις δύσκολες συζητήσεις. Να μην τις κρύβουμε κάτω από το χαλί. Όντως, έχουμε την πρόκληση μεγάλη της ζωσπαστικοποίησης των νέων. Όλοι οι δάσκαλοι περνάνε από αυτό. Αλλά και εμείς ως πολιτικοί έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. υπουργοί. Άρα λοιπόν πρέπει να συζητάμε μεταξύ μας και για δύσκολα θέματα. Και θα το κάνουμε. Καταπολέμηση των ανισοτήτων τώρα όπως ρώτησε και η κυρία Βάρτ, όντως θέλουμε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Θέλουμε ένα, μια θετική νότα εδώ και συμφωνώ μαζί σας με τη θετική προσέγγιση δηλαδή που έχετε απέναντι στους νέους πράγματι. Υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι με ιδεώδη, με ιδέες και αυτούς πρέπει να τους προσεγγίσουμε. βρίσκονται στην Ευρώπη και πρέπει να φτάσουμε εμείς αυτούς. Πρέπει επίση, και όντω και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα επανέλθει ξανά και ξανά στο Συμβούλιο, η ριζοσπαστικοποίηση όπως είπα και πριν που δεν θέλουμε να το κρύβουμε το θέμα κάτω από το χαλί και η κυρία άλλοι ρώτησαν. Ναι, όντω η θέση των γυναικών και η άποψη των γυναικών πρέπει να ακούγεται. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα αυτό. Και το καλό παράδειγμα είναι ακριβώ αυτό που θα ζητήσω από τους συναδέρφους. Και αυτό να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ συνεργάζομαι με τον συνάδελφο Φαν Θα σας απευθύνει και αυτό το λόγο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία μας. Πρώτα λοιπόν εγώ κοιτάω την εκπαίδευση, τη δήλωση του Παρισιού που έκαναν οι Υπουργοί Εκπαίδευσης, αλλά μερικά θέματα πάνε και πέρα από το σχολείο. Έχουν να κάνουν με θεσμούς τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν οι γονείς, οι άλλοι κοινωνικοί παράγοντες. Για τον κύριο Διακόνα, η εκπαίδευση φυσικά είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Δεν φτάνει όμως από μόνη της. Ούτε μπορούμε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας να στήσουμε από τους δασκάλους να τα λύσουν. Όχι, πρέπει και εμείς να σκεφτούμε πώς με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας, ε, γνωρίζοντας ε, καλύτερα ποιος έχει πια αρμοδιότητα στην εκπαίδευση, να αναλάβουμε και εμείς μέρος των αρμοδιοτήτων που έχουν οι δάσκαλοι ή να τους στηρίξουμε στις δικές τους αρμοδιότητες. Και αυτό πώς θα γίνει, θα γίνει αν συζητήσουμε με κοινωνικούς λειτουργούς που ασχολούνται με τους νέους, ακόμα και με θρησκευτικέ οργανώσεις, όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον περίγυρο των νέων. και στην κυρία Φένερα, αν λέω καλά το όνομά τη, λέει υπουργό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διαφορές, τις πολιτισμικές, να δούμε ποιες είναι οι αρχές της Ευρώπης, τι γίνεται με τη διαπολιτισμικότητα και την ένταξη των ξένων. Στην κυρία Χιμένες που ρώτησε τι κάνουμε με τα ρεύματα τα μεταναστευτικά. Σα είπα και πριν, δεν τα κρύβουμε κάτω από το χαλί αυτά τα θέματα, παρόλο που είναι δύσκολα. Γιατί πολλέ φορέ αποτελούν και πηγή νέων ιδεών υπέρ τη πολυπολιτισμική διαδικασία. Όπως και να έχει το πράγμα πάντω, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κοινωνικές επαφές και να ενισχυθούν αυτές ανάμεσα στους μετανάστες και τον τόπιο πληθυσμό για να δημιουργηθούν δεσμοί και γι' αυτό θέλουμε τον πολυπολιτισμικό διάλογο και αποτελεί προτεραιότητα στο Συμβούλιο αλλά και στη... είναι προτεραιότητα και της Ολλανδικής Προεδρίας για το εξάμεινο αυτό και για τις δύο επόμενες προεδρίες, για το τρίο των προεδρών δηλαδή για τον πολιτισμό. Η κυρία Κάμερετ και ο κ. Μοργάνο με ρωτήσατε για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Αυτό που μπορώ να σας απαντήσω τώρα, τι θα κάνει η Ολλανδία δηλαδή, είναι ότι το Νοέμβριο το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να κάνει την πρόταση για το έτος αυτό. Και από ό,τι κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει πρώτα, οπότε την περιμένουμε, αν αποφασιστεί να υπάρξει ένα τέτοιο έτος, ευρωπαϊκό δηλαδή, τότε πιστεύω ότι ο πολιτισμός, η πολιτισμική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ένα καλό θέμα και αυτό θα ζητήσουμε κι εμείς. Έρχομαι τώρα στην Ευρωπαϊκή. Πολύ χαίρομαι που ακούω το ενδιαφέρον σας που με ρωτήσατε για το Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Σόντροβα για την παρατήρησή της όσον αφορά την στήριξη της τσεχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή. Όντω έχω μιλήσει πολλούς από την Ευρωπαϊκή και έχω την αίσθηση ότι τώρα κάτι πρέπει να γίνει όσον αφορά την Ευρωπαϊκή. Αν δεν κάνουμε τώρα τίποτα, τότε θα χάσουμε την ευκαιρία και θα χάσουμε και αυτό που ήδη έχουμε. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας και την ενθάρρυνσή σας και την κυρία Τρίπελ και τον κύριο Σοτροσκεύσκη. Αν προφέρω πάλι καλά το όνομα. Ναι. Όσον αφορά την χρηματοδότηση και την ε, προβολή της Ευρωπαϊκής αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και σε επίπεδο χωρών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου στα συμπεράσματα του Συμβουλίου να αναφέρεται κάτι γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή πρέπει όντω να προβληθεί περισσότερο και να γίνει περισσότερο γνωστή στους Ευρωπαίους πολίτες υπάρχει όντω ένα πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι κάτι που μπορεί να προωθηθεί και θα έπρεπε να προωθηθεί περισσότερο. Στον κύριο και όσον αφορά το πολιτιστικό πρόγραμμα της Ολλανδίας. Ναι, έχουμε και στις Βρυξέλλες και στο Άμστερνταμ και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στο κτίριο της Ευρώπης στο Άμστερνταμ θα λάβουν χώρα πολλές συναντήσεις Ολλανδοί σχεδιαστές και καλλιτέχνες έχουν δραστηριοποιηθεί και σας προσκαλώ όλους από βάθους καρδιάς να έρθετε για να δείτε αυτά τα δημιουργήματα. Να δείτε δηλαδή τι έχει να προσφέρει η Ολλανδία πολιτιστικά. Παρόλο βέβαια που βρισκόμαστε σε περιόδους οικονομικής κρίσης και σφιξίματος, παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά και εμείς θέλουμε, όπως σας είπα και σε διεθνές και σε διεθνές επίπεδο, την επαφή αυτή μέσω της εκπαίδευσης με τους νέους και τους λιγότερο νέους. Σας εύχομαι λοιπόν και σας καρποφόρες εργασίες. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι δεν είμαι σε θέση να απαντήσω ίσως πολύ συγκεκριμένες όλες σας τις ερωτήσεις, αλλά βρισκόμαστε μόνο στην αρχή του διαλόγου μας. Έχουμε ένα εξάμεινο για να μπορούμε να συζητάμε μαζί. Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πρέπει να προωθούνται γιατί προωθούν και αυτά τα ίδια τις ευρωπαϊκές αξίες. Ο πολιτισμός περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οπότε ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Θα χρησιμοποιήσω τα σχόλιά σας, θα τα κρατήσω. Και θα προσπαθήσω να προχωρήσω περισσότερο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού στο Συμβούλιο για να μπορέσω να έχω και περισσότερο να σας πω την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, για την ομιλία σας και τις δεσμεύσεις που αναλάβατε. Πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και συντονίζονται με τις ευαισθησίες και τις προτάσεις Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Θα ήθελα να αποστείλω ένα τελευταίο μήνυμα, μικρό μήνυμα που αφορά την ένταξη και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Εδώ στο Κοινοβούλιο ψηφίσαμε μια σημαντικότατη έκθεση για την υποστήριξη της πρόσβασης των παιδιών και των νέων προσφύγων στην παιδεία, των προσφύγων στα στατόπεδα των προσφύγων. 23 εκατομμύρια περισσότερα πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε το ποσό να διπλασιαστεί, αλλά και να έχουμε και τα ελάχιστα, ελάχιστε προδιαγραφέ στην υπόδοχη τη χώρα μα. Χρειάζεται μια δέσμευση από αυτό. Και άλλη πρόταση που κάναμε ήταν να δημιουργηθεί ένα διάδρομο εκπαιδευτικό, τον αποκαλέσαμε έτσι, για τόσα παιδιά ε, από τη Συρία και άλλες, ε, από άλλες χώρες που ζήτησαν να έρθουν στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ζητήσαμε υπάρχει διαθεσιμότητα από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και, και τα μαθήματα εξ αποστάσεως επίσης να έχουν, ε, να έχουν πρόσβαση. Συζητήσαμε ε, στην Επιτροπή μαζί με τις διμερείς αντιπροσωπείες διαφόρων χωρών, τρίτων χωρών, το συζητήσαμε. Θα ήταν καλό στο Συμβούλιο επί Ολλανδικής Προεδρίας που είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό να υπάρξει υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση και στα συγκεκριμένα αιτήματα, ερωτήματα που, για την πολιτισμική κληρονομιά για το Ευρωπαϊκό Έτος του 2018 και τα αιτήματα που ευλήθησαν έστειλε στον Διπρόεδρο Τίμερμας που τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά μια επιστολή. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε πάρει απάντηση ικανοποιητική. Σίγουρα πιστεύω ότι η Προεδρία σα θα είναι στατική σημασία, όπω αναφέρατε και πριν, προ αυτή την κατεύθυνση. Διότι αν το αποφασίσουμε τώρα θα είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Υπάρχει μεγάλη προσοχή στον κόσμο τον πολιτισμικό από τη δημιουργική βιομηχανία, την πολιτισμική. Θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα πολύ ισχυρό που κινδυνεύει να χάσει την πολιτισμική της ε, διάσταση και τη διάσταση αλληλεγγύης. Θα σας χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε και βασίζομαι πάρα πολύ στη συνεργασία μαζί σας και στο Συμβούλιο. Ε, Κυρία Υπουργό, να δώσω μια απάντηση στις ερωτήσεις σας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Για μένα προσβλέπω στις πληροφορίες που έχετε σαν Επιτροπή και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές στα βήματα που θα κάνουμε. Επίσης θα διοργανώσουμε μια διάσκεψη και μια άτυπη συνάντηση ε, στο διαδίκτυο για την ανοιχτή εκπαίδευση ε, εξ που κυρίως είναι ε, για ανώτατη εκπαίδευση αλλά μπορεί και για τη διαβίου εκπαίδευση χρησιμοποιείται και την εκπαίδευση των ηλικιωμένων αλλά επίσης και για την εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστών. Ε, ξέρετε, έχουμε επίγνωση αυτής της δυνατότητας και θα δώσουμε τη δέουσα προσοχή και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Κώστα. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Και τώρα, κύριε Υπουργέ Αθλητισμού, Υγεία, ε, Υγείας και Ευημερίας, Μάρτι Βαν Ράιεν, δεν ξέρω να προφέρω σωστά το όνομά σας, αν έχετε την καλοσύνη να έρθετε να καθίσετε εδώ. Okay, okay. And so, the change of the church. Συνάδελφοι, μόλις μισή ώρα έχουμε για την ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον αθλητισμό. Ελπίζω να μείνετε για να ακούσουμε τον κύριο Υπουργό. Αν με επιτρέπετε θα συνεχίσω τελικά, θα ήθελα να πω απλώς αυτό ότι έχουμε τον Υφυπουργό Υγείας, Αθλητισμού και Ευημερίας και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι καλύπτει αυτές τις αρμοδιότητες. Σίγουρα αυτές οι διαστάσεις του αθλητισμού και της παιδείας είναι πάντα παρόντα εδώ. Η Ολλανδική Προεδρία γνωρίζω ότι ήδη προέβλεψε σημαντική εκδήλωση στη Χάγη τον Μάρτιο αλλά δυστυχώ με το Ευρωπαϊκό Φόρουμο του Αθλητισμού, ακριβώ όταν εμεί θα έχουμε την Ολομέλεια στο Στρασβούργο, αυτό είναι ένα θέμα που δυστυχώς για μας ε, δημιουργεί πρόβλημα. Κάθε φορά που εμείς δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε, διότι είμαστε στην Ολομέλεια, φοβάμαι ότι λίγοι συνάδελφοι θα μπορέσουν να παραστούν, αλλά σίγουρα ενδιαφερόμαστε για τα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός, η αθλητική πρακτική και η εκπαίδευση για τον αθλητισμό και η παιδεία των αθλητισμών σαν είδο τρόπο ζωής και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας είναι ένα θεμελιώδες θέμα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, ε, και το πώς παρουσιάσατε στην Ολλανδική Προεδρία την ακαιρεότητα και τη διαφάνεια στον αθλητισμό και πόσο μεγάλες συνέπειες μπορούν, να αντίκτυπο έχουν οι μεγάλες θετικές εκδηλώσεις και οι μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούν οι θετικές εκδηλώσεις, ούτως ώστε να αναπτύσσεται και αυτή η διάσταση. Ε, έχει και οικονομικό αντίκτυπο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, μας ενδιαφέρει να επικρατεί η διαφάνεια εκεί που διοργανώνονται εκδηλώσεις, όπως υπογραμμίσαμε ήδη. Και με την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας ενδιαφέρει όσον αφορά την επιλογή των τόπων, τοποθεσιών που γίνονται μεγάλες θετικέ εκδηλώσεις και να μην επηρεάζουν τα οικονομικά πάνω απ' όλα την επιλογή. Λοιπόν, σα δίνω το λόγο και σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας και μετά θα είμαστε όλοι πολύ συνοπτικοί σε ερωτήσει που θα υποβάλλουμε. Λοιπόν, έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω το θεματολόγια και τις προτεραιότητες του δομέα και του αθλητισμού επί Ολλανδικής Προεδρίας. Όπως συζητήσατε, Υποστήκαμε όλοι σοκ τον τελευταίο Νοέμβριο από τις επιθέσεις ε, στην, στο Παρίσι, δέκα μόλις μήνες μετά τις αντίστοιχες επιθέσεις στο Σαρλί Και το ζήσαμε και στις ε, Βρυξέλλες εδώ, στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, ε, που έχει καλυφθεί από σώματα ασφαλείας λόγω των σοβαρών και επικείμενων απειλών για επιθέσεις όλοι μας ε, ε, ανησυχούμε για την ε, άνοδο του ISIS και του βίου εξτρεμισμού. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να καταπολεμήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Έχουν ήδη αναλυφθεί διάφορες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν τα πιεστικά αυτά προβλήματα. Ωστόσο χρειαζόμαστε και μια πακροπρόθεσμη λύση και οι σημαντικότερες λέξεις έννοιες ε, σε αυτό το τομέα είναι η έννοια της πρόληψη. Χρειαζόμαστε ασφάλεια και δικαιοσύνη για την πρόληψη των επιθέσεων. Χρειαζόμαστε ε, πρόληψη του βιοεξτρεμισμού αλλά θα πρέπει να προλαμβάνουμε και την ίδια τη ριζοσπαστικοποίηση. Γι' αυτόν τον λόγο η ριζοσπαστικοποίηση ή, να το πω καλύτερα, η πρόληψη του βιοεξτρεμισμού μας αφορά όλους και βρίσκεται πάνω-πάνω στην ατζέντα μας. Τα πρόσφατα γεγονότα τονίζουν ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, όχι μόνο όσον αφορά την πολιτική ασφάλεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και δικαιοσύνη, αλλά και όσον αφορά την ένταξη, την κοινωνική ένταξη νέων ανθρώπων, καθώ η ριζοσπαστικοποίηση πολύ συχνά ε, ξεκινά σε πολύ μικρή ηλικία. Η Ολλανδική Προεδρία θα ήθελε να δώσει στην πρόληψη την ε, προσοχή που χρειάζεται όσον αφορά την πρόληψη δηλαδή της ριζοσβαστικοποίησης. Η ζωσβαστικοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε βιοεξτρομισμό και είναι ένα πρόβλημα που αφορά νέους ανθρώπους από διάφορα πολιτικά περιβάλλοντα. Θεωρούμε ότι οι νέοι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την πρόληψη του βιοεξτρεμισμού. Όπως αναφέρεται στην κοινή έκθεση του Συμβουλίου και τη Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του επικαιροποιημένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα τη νεολαία, απαιτείται μια διατομιακή ε, προσέγγιση. Απαιτείται μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων για να μεγαλώσει κάνει ένα παιδί, αλλά χρειάζεται και μια κοινότητα ανθρώπων για να προλαμβάνεται η πριζοσπαστικοποίηση των νέων και η ε, ε είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι δηλαδή να θεωρούν ότι είναι τμήμα της κοινωνίας. Στη διάρκεια της Λουξεμβουργικής Προεδρίας συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι δραστηριότητες για, για τους νέους για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εκεί όπου ζουν οι νέοι άνθρωποι η κοινωνική λειτουργή μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον προσδιορισμό της ταυτότητας των νέων ανθρώπων. Οι δραστηριότητε για τους νέους, ο εθελοντισμός, ο αθλητισμός, οι πολιτικές δραστηριότητε μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία για να απευθυνθούμε στους νέους ανθρώπους. Αυτά τα εργαλεία αυτής της πολιτικής μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ανθρώπους, νέους ανθρώπους, του οποίους κανονικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πολύ συχνά η... το ISIS χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να στρατολογήσει νέους ανθρώπους. Εμείς χρειάζεται και οι κοινωνικοί λειτουργοί μας να μπορούν να δραστηριοποιούνται και, και εκείνοι ε, στο, διαδίκτυο. Διότι άπαξ και δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών λειτουργών με τους νέους ανθρώπους μπορούν να τους καθοδηγήσουν όσον αφορά την, τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους. Κάτι που ε, είναι απαραίτητο. Οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται μια αίσθηση του ανήκει, μια αίσθηση της συμμετοχής για να μην είναι ευάλωτοι σε ριζοσπαστικές επιρροές και θα πρέπει να, να ενισχυθεί η, συνεργασία μεταξύ σχολείων, εκκλησιών, ε, γονέων, τζαμιών. Σε συνεργασία με την ε, συνάδελφο υπουργό με την οποία μιλήσατε λίγο νωρίτερα, θέλουμε να ε, αναπτύξουμε μια προσέγγιση διατομεακή και να καταλήξουμε σε μια κοινή στάση όσον αφορά την αντιμετώπιση της ζωοστικοποίησης. Και εμείς θα θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά την ε, διερεύνηση διαφόρων δυνατοτήτων που έχουμε και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διακήρυξη για την προώθηση της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών για τις ελευθερίες αντοχής και της μη διάκρισης που υπαγράφει από τους Υπουργούς Παιδείας τον Μάρτιο του 2015. Αυτή η διακήρυξη αποτελεί τη βάση της διατομιακής προσέγγισης και παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τον τρόπο συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση και για την προώθηση τη ιδιότητα των πολίτων μεταξύ των νέων ανθρώπων. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε εμπειρίε σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίε μπορούν να ανταλλαχθούν. Διότι διακυβεύεται το μέλλον τη Ευρώπη. Αυτό το γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και γιατί ακριβώ παλεύουμε. Φυσικά η πρόληψη του βίου χρειάζεται περισσότερα πράγματα. Εργασία, απασχόληση, εκπαίδευση, η ασφάλεια και η πολιτική για την νεολαία είναι σημαντική τομή, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζουν. Και εμεί προσβλέπουμε προ τη συνεργασία μαζί σα και με όλου του εμπλεκόμενου φορεί για, να για να μπορέσουμε να δούμε πώ θα, θα μπορούσαμε να προλάβουμε τον βίαιο εξτρεμισμό. Εμείς θα καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και την περιοθεροποίηση των νέων ανθρώπων με σκοπό να καταλήξουμε και συμπεράσματα συμβουλίου για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης με σκοπό να υιοθετηθούν τα συμπεράσματα αυτά στο Συμβούλιο Παιδείας Νεολαίας Πολιτισμού και Αθλητισμού τον Μάιο του 2016. Το ίδιο θέμα θα συζητηθεί και στο συνέδριο που θα διοργανίσουμε ε, με στις 17 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μάστρη σχετικά με την ψυχική υγεία των νέων. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο διαστρωμένο διάλογο. Όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να, νιώθουν ότι είναι τμήμα της κοινωνίας. Και αυτό βεβαίως ισχύει για όλους τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό οι φορείς χάραξης πολιτικής να έχουν στενή σχέση με τους νέους αυτούς ανθρώπους. Η Ολλανδική Προεδρία θεωρεί ότι ο διαστρωμένος διάλογος είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ε, για την, ε, <clears throat> από τα κάτω προς τα πάνω για να συνδεθούμε με τους νέους ανθρώπους. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μάθουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση την οποία βιώνουν οι νέοι άνθρωποι. Και στο πλαίσιο του διαδρομένου διαλόγου, το τρίο προεδριών μεταξύ κάτω χωρών ε, Σλοβακίας και Μάλτα θα εργαστεί προκειμένου να, να καταλήξουμε σε μια θεματική προτεραιότητα για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 16 έως 30 Ιουνίου 2017 και ο, ο τίτλος θα είναι δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν με πολύμορφο και συνδεδεμένο τρόπο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτοιμοι για τη ζωή, έτοιμοι για την κοινωνία. Σε αυτή τη διάρκεια, σε τη διάρκεια αυτών των 18 μηνών θα διοργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις και το κύριο ε, συμβάν επί Ολλανδικής Προεδρίας είναι ε, το, το, η συνδιάσκεψη για την νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διοργανωθεί 5-7 Απριλίου 2016 στο Άμστερνταμ. Να περάσω και στον αθλητισμό. Καταρχάς να πω δύο λόγια για το στήσιμο των αγώνων. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα εκκρεμές ζήτημα στον τομέα του αθλητισμού που είναι η υπογραφή του, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το στήσιμο αγώνων. Δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν επί Λουξεμβουριανής και Λετωνικής Προεδρίας παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Η Προεδρία θα προσπαθήσει να εξετάσει πώς θα μπορούσαν να προωθηθούν αυτές οι προτάσεις στο Συμβούλιο. Η Ολλανδική Προεδρία έχει σκοπό να οργανώσει ένα, μια συνάντηση με το Συμβούλιο της Ευρώπης και να διευκολύνει ε, τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν, να υπογράψουν την σύμβαση αυτή. Θα πρέπει στο, ε, στην περίοδο 2014-2017 να ενισχύσουμε το ζήτημα της ακεραιότητας του αθλητισμού. Αυτό το ζήτημα το έχετε δείξει και εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Όπως γνωρίζετε, ο αθλητισμός αντιπροσωπεύει πολλές θετικές αξίες όπως είναι η ευχαρίστηση, η περηφάνεια, οι επιδόσεις και η συνεισφορά του στην ευμερία και την υγεία δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Γι' αυτόν τον λόγο η ακαιρεότητα, η διαφάνεια και η καλή διακυβέρνηση είναι σημαντικότατοι παράγοντε και εργαλεία στην πρόθεση του αθλητισμού. Ω κυβερνητικέ οργανώσει μπορούμε να υποστηρίξουμε το κίνημα του αθλητισμού ε, ω προ την απαραίτητη διαδικασία για την ε, δημοκρατική και οικονομική ευγενή άμυλα. Μπορούμε να καταλήξουμε συμφωνίε όσον αφορά την ε, σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών για την καλή διακυβέρνηση την ε, ακεραιότητα και την ε, διαφάνεια. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η ανάληψη των καθηκόντων ε, από την πλευρά του Τόμας Μπαχ, των καθηκόντων του ως Προέδρου του της ΔΟΕ. Θεωρούμε ότι η Ολυμπιακή Ατζέντα 2020 ενστερνίζεται τις αξίες και τις αρχές για τις οποίες παλεύουμε και εμείς θεωρούμε ότι μια κοινή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε ε, προστιθέμενη αξία για την προώθηση για την, ε, τις ε, τι της και της καλής διακυβέρνησης στις μεγα... και για τον αθλητισμό γενικά αλλά και για τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και για το στόχο αυτό η Ολλανδική Προεδρία θα ε, επιδιώξει να ε, εκδοθεί μια πολιτική δήλωση σχετικά με την ε, ακαιρεότητα στον αθλητισμό. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και συμπεράσματα συμβολή σε συνεργασία με τον κόσμο του αθλητισμού. Τα παραδοτέα των ομάδων εμπειρογνωμόνων αφορούν την καλή διακυβέρνηση και την οικονομική αξία του αθλητισμού. Θα προσπαθήσουμε να τα συμπεριλάβουμε στα, συμπεράσματα. Για το αντι doping Τα τελευταία χρόνια ε, είχαμε διάφορα σκάνδαλα ντόπινγκ και, στην, ε, και στο στίβο αλλά και στην ποδολασία και αλλού. Είναι πολύ σημαντικό στον τομέα του αντι-doping η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ισχυρή φωνή. Η Ολλανδική Προεδρία θα προετοιμάσει συντονισμένες ευρωπαϊκές θέσει σε σχέση με το έργο που βρίσκεται εξέλιξη στη Γουάντα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, οι ευρωπαϊκές θέσεις θα παρουσιαστούν από τους τρεις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο, στις συναντήσεις της ΟΑΝΤΑ το Μάιο του 2016. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε, να βεβαιώσουμε μάλλον τη ΟΑΝΤΑ ότι ο νέος κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στο έργο του anti-doping. Εμείς ως Ολλανδική Προεδρία θα διοργανώσουμε και ένα σχετικό συνέδριο όπου θα προσπαθήσουμε να, ε, να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα ντόπινγκ και να καταδείξουμε και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο νέο κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, στις 9 και 10 Μαρτίου 2016 θα γίνει το Φόρουμ Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χάγη της Ολλανδίας. Το φόρουμ αυτό οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή μου έχει υποσχεθεί ότι θα προσκληθούν στο φόρουμ αυτό και ευρωβουλευτές. Στις 10 και 11 Μαρτίου, έπειτα από το Φόρμα Αθλητισμού, θα ε, ε, γίνει ε, η συνάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού και το Συμβούλιο Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί 31 Μαΐου 2016. Την ίδια μέρα μάλιστα θα γίνει και διαρθρωμένος διάλογος στις Βρυξέλλες. Και τέλος θα διοργανώσουμε και ένα συνέδριο κατά του ντόπινγκ στο Άμστερνταμ του του, του 15 Ιουνίου του 2016. Ένα τελευταίο μήνυμα. Ο αθλητισμό είναι χαρά, αλλά αυτό ισχύει μόνο αν χαρακτηρίζεται από ευγενή άμυλα. Άρα η ακαιρεότητα, η διαφάνεια και η καλή διακυβέρνηση μπορεί να επαναφέρουν τον αθλητισμό στι βασικέ του λειτουργίες, στις βασικές του λειτουργίε, για το άτομο αλλά και για την κοινωνία ω σύνολο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρέμβασή ε, Υπήρξα ακούγεται ακριβέστατος επί κάποιων θεμάτων. Άκρο ενδιαφέρουσε υποχρεώσει υποχρεώσεις που αναλάβατε για την Ολλανδική Προεδρία. Τα τρία θέματα αυτά που αναφέρατε μας απασχολούν πολύ, δηλαδή ότι ο αθλητισμός είναι ένα μεγάλο εργαλείο ένταξης και πρόληψης τη ζωστικοποίησης και χρειάζεται η ενεργή συμμετοχή των νέων που μπορούν να συμμετέχουν και αισθάνονται ανήκουν. δημιουργούν μια ταυτότητα θετική λοιπόν. Ε, το ότι αναφερθήκατε για την πολιτική δήλωση μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για την ακαιρεότητα του αθλητισμού είναι κάτι που το συμμεριζόμαστε. Νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό. Και το άλλο που θίξατε για την σύμβαση αυτή για το να μην στείνονται τα, οι αγώνες. Λοιπόν, θα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει αυτή την τη σύμβαση. Ελπίζω να επαναπροθεθεί όλη η ε, πρωτοβουλία. Και τέλος σημαντικότατη υποχρέωση για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, συμμετάσχουμε στο συνέδριο, αλλά είναι η τελευταία ημέρα του Στρασβούργου με τις ψηφοφορίες. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο τρόπο, ώστε αν και υπάρχει αυτό το εμπόδιο και δεν υπάρχει ο συντονισμό, να καταφέρουμε να έχουμε κάποια παρουσία του Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο αμέσω σε εκείνου που ζήτησαν το λόγο. Ουέντα, για δύο λεπτά αντιπρόεδρος και εθνικός πρωταθλητής του handball. Οπότε γνωρίζει καλά το, το θέμα, ξέρει τα θέματα του αθλητισμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτά που μας είπατε. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί και χαίρομαι διότι μετά μερικά από αυτά που είπατε στην παρουσίασή σας όπως το ντόπινγκ, το στήσιμο των αγώνων ή ε, η ανάθεση διαφόρων ε, αθλητικών ε, εκδηλώσεων είναι πρόβλημα. Η εκλογή του Τόμας Μπαχ ήταν ένα καλό βήμα. Θα ήθελα να πω ότι δημιουργήσαμε μια διακοινοβουλευτική ομάδα για τον αθλητισμό. Είναι νέα ομάδα, για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Εγώ ε, είμαι αναμεμειγμένος πολύ με τον αθλητισμό, αλλά θα ήθελα να κινηθώ σε κάτι άλλο επίσης που αναφέρατε, την κοινωνική ένταξη, κυρίως την ένταξη των μεταναστών διοργανώσαμε μία συνάντηση με διάφορα κόμματα και διάφορους, διάφορα μέλη. Ένας νέος Αφγανός πρόσφυγας πήρε το λόγο εκεί σε αυτή την εκδήλωση και είπε ότι ο αθλητισμός τον βοήθησε να δημιουργήσει κοινωνικές δραστηριότητες, τον βοήθησε να ενταχθεί. Αισθάνθηκε ότι έγινε αποδεκτός. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό μας δείχνει την κατεύθυνση που αναφέρατε και εσείς, την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε. Ότι ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας να πετύχει και άλλους στόχους ο αθλητισμός. Το επόμενο που έχω να πω είναι η FIFA και η UEFA. Διοργανώνουμε συναντήσεις με τους επικεφαλείς των φορέων αυτών διότι πιστεύω ότι μπορούμε να δείξουμε πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Μετά από αυτή την ιστορία των σκανδάλων μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Θα πρέπει να ενώνει αθλητισμός, να είναι συνδετικός συστός. Όχι μόνο να συνδέει κοινωνικά τους ανθρώπους, αλλά είναι σημαντικός αθλητισμός και για την οικονομία. Δεν είναι θέμα συναισθηματικής συμμετοχής αποκλειστικά, όπως είπε η κυρία Κώστα, και αλλά έχει και άλλα στοιχεία. Το, το, το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Ουκρανία και την Πολωνία το 2012, το ευρώ. Ε, πολλοί τουρίστες ε, ήρθαν στην Πολωνία και αυτό δείχνει ότι μέσω του αθλητισμού έρχονται τουρίστες και γνωρίζουν τη χώρα και μαθαίνουν τις χώρες. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Η Έλγα Τρούπελ έχει το λόγο. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομο. Γιατί είμαστε, μας τελειώνει ο χρόνος για τους νέους. Of... Και φαστικοποίηση ή αποφυγή φαστικοποίησης. Να δώσω ένα παράδειγμα από τη Γερμανία. Uh, Έχουμε έναν Άραβα Ισραηλινό που είναι ψυχολόγος στη Γερμανία και εργάζεται με νέους για να αποφύγει τη φαστικοποίηση ή να απορριζαστικοποιεί. Και νομίζω ότι αυτά που είπατε στηρίζουν αυτά που μας είπε. Πρέπει να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές, τα παραδείγματα διαφόρων κατών μελών. Να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να δούμε τι καλύτερο κάναμε τελευταία χρόνια. Και να αποφύγουμε τελικά να φεύγουν οι νέοι και να πηγαίνουν στο τζιχάντ. Συνάδελφε Μπόξκορ, αντιπρόεδρε της Επιτροπής, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Θέλω να αναφερθώ λίγο στην στρατηγική 2013-2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ετοιμάσω με αυτό το αντικείμενο μία έκθεση. Οπότε και εγώ θέλω να ρωτήσω για τους νέους, για την Ευρωπαϊκή Νολέα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι η νεολαία αποτελεί προτεραιότητα για την Προεδρία σας. Και χαίρομαι επίσης που άκουσα ότι θα επικεντρωθείτε πολύ στους νέους της κοινωνίας μας. Επίσης η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό θέμα προκειμένου όλοι οι νέοι να έχουν θέση στην αγορά εργασίας. Άρα πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες, δυνατότητες στους νέους από αυτού. Και χάρηκα που σας άκουσα να λέτε ότι οι τοπικές κοινότητες έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και η οικογένεια, οι θρησκευτικέ κοινότητες, οι εκκλησίες όπου πηγαίνουν οι νέοι κλπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ρόλο προκειμένου να προετοιμάσουν τους νέους για το μέλλον και να εμποδίσουν ακριβώ αυτούς τους νέους να στραφούν προς εξτρεμιστικές οργανώσεις. Άρα οι τοπικές κοινότητες και ε, τα σχολεία ή οι οργανώσεις όπου πηγαίνουν οι νέοι σε τοπικό επίπεδο έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Τώρα το θέμα των μειωτικών γλωσσών και του δικαιώματος πρόσβασης στον ε, πολιτισμό μικρών κοινοτήτων, μειονοτήτων. Θα πρέπει όλοι να μπορούν να έχουν τέτοια πρόσβαση. Πρέπει και να εντάσσονται στις κοινωνίες μας, αλλά να εξακολουθούν να έχουν σχέσεις με τις δικές τους κοινωνίες στη χώρα τους. Έχουν έρθει τελευταία πολλοί και έχουν βρεθεί με άλλους που έχουν έρθει από παλιότερα στις χώρες μας. Όλα αυτά βοηθούν στην πολυπολιτισμικότητα της Ευρώπης. Όλα αυτά για να σας ρωτήσω και το εξή τελικά. Τι θα κάνετε για να μειωθεί η ανεργία των νέων, τι θα κάνετε για να βοηθήσετε τους νέους με τον αθλητισμό ή μέσω του αθλητισμού. Ευχαριστώ και εδώ θα δώσω το λόγο για την απάντησή του. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για να απαντήσω στον κύριο Ρέντα, ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία που ανέλαβε η ε, κοινοβουλευτική αυτή και κοινοβουλευτική αυτή ομάδα για τον αθλητισμό και 24 Νοεμβρίου έφτασε στο Νοέμβριο ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις βέλτιστες πρακτικές της χώρες μέλη έδειξαν ενδιαφέρον οι χώρες πώς να χρησιμοποιήσουν δηλαδή τον αθλητισμό υπέρ των νέων και για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες να μπορούν και αυτοί να έχουν πρόσβαση στον Η Προεδρία μας γνωρίζει επίσης την ε, πρωτοβουλία που θα έχουμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα συμπεριλάβει την νεολαία και έτσι θα δούμε ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα. Το παράδειγμα που δώσατε με εξέπληξε εκείνου του Αφρικανού είπατε που είπε ότι δεν επρόκειτο μόνο για θέμα πολιτισμού ή για κάτι που κάνει κανείς μόνος του, είναι μια κοινωνική δραστηριότητα. Είναι εντυπωσιακή αυτή ιστορία. Μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Και είναι καλό να τις χρησιμοποιούμε και στη χάραξη πολιτικής μας. Όντως, να χρησιμοποιήσουμε τον αθλητισμό σαν μέσο ένταξης. Στην κυρία Τρούπελ τώρα θέλω να απαντήσω. Ευχαριστώ που προθείτε αυτό που φαίνεται να είναι Πολύ καλό βιβλίο, πώς να το διαβάσω. Είναι σημαντικό, αν το συζητήσω, το θέμα της ένταξης με τους συναδέρφους μου, πάντα διαπιστώνω ότι είναι δύσκολο να χαράξει κανείς πολιτική λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση αυτή της ένταξης και σε εθνικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα. Πόσο μάλλον σε διεθνές επίπεδο. Αξίζει όμως τον κόπο. ίσως να μην παίζει τον αποφασιστικό ρόλο στην ένταξη, αλλά αν δεν χρησιμοποιήσουμε τέτοιες ευκαιρίες, δεν θα έχουμε και επιτυχία. Δύσκολη εφαρμογή. Όλες μας οι χώρες το συζητούν σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές μεταξύ μας. Με την κυρία Φόξερ τώρα. Ευχαριστώ για την στήριξή σας στις προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας. Όντως αυτή η δύναμη των τοπικών κοινοτήτων μπορεί να βοηθήσει στην ίδια την ανάπτυξή τους και μία από τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε στην Ευρώπη είναι να μην έχουμε ένα είδος πολιτισμού, να έχουμε πολλαπλές μορφές πολιτισμού. Πολύ σημαντικό λοιπόν να το πάμε ακόμα πιο μακριά. Για την ανεργία, προωθούμε τις, τις δεξιότητες και είναι κάτι που προωθούμε στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να είναι μέρος και αυτής της ολοκληρωμένης πολιτικής. Δεν πρέπει δηλαδή να συνεργαζόμαστε μόνο μεταξύ Υπουργών ε, Νεολαίας και τα λοιπά, αλλά και με τους Υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλους που είναι αρμόδιοι για τις πολιτικές απασχόλησεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη στήριξή σας και προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί για να προχωρήσουμε αυτό το θέμα ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πραγματικά κύριε Υπουργέ, ίσως τα... ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Να πω αυτό υπό το φως αυτών που είπαν οι συνάδελφοι και εκείνων που εσείς υπενθυμίσατε πριν, δηλαδή μετά τη δήλωση των Παρισίων τι γίνεται. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν έχουμε χρόνο, να ακούσουμε και εκπρόσωπο την ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίαση που θα έχουμε τον Επίτροπο Ναύρασίτς μετά την δήλωση των Υπουργών στο Παρίσι θα είναι σημαντικό να αναλυθεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει ακριβώς ολιστικά και εγκάρσει όλα τα θέματα που περιγράψατε. Όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε στην παιδεία, εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, προσπάθειες για ένταξη. Χρειάζεται μια απάντηση πολιτική Διαφορετικά θα περιθωριοποιηθεί το θέμα αυτό σε σχέση με τα πλήρη προγράμματα. Μπορούμε να βασιστούμε στην Ολλανδική Προεδρία, θα μας στηρίξει έτσι, όπως είπε και η Υπουργό Παιδείας και όπως είπατε τώρα και χαιρόμαστε για τις υποχρεώσεις που αναλάβατε, τις δεσμεύσεις που αναλάβατε. Γι' αυτό ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και θα τα ξαναπούμε ελπίζω να τα πούμε και στις 10 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, λοιπόν, η επόμενη συνεδρίαση, Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου. Τετάρτη και Πέμπτη, 18 του μηνός, από τις 9 μέχρι τις 12.30. Προηγούμενη μέρα ολόκληρη Τετάρτη. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς την Πρόεδρο. και όσοι αποχωρούν από την αίθουσα ας αποχωρήσουν γρήγορα παρακαλώ διότι έχουμε καθυστερήσει και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε όσοι δεν έχουν σχέση με αυτή τη συνεδρίαση παρακαλώ θερμά να αποχωρήσουν.